Einen schönen guten Καλημέρα σας. Άρχεται η συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα κάποιες ανακοινώσεις. Οι αρχές της Λετωνίας υπέβαλαν έτοιμα άρσης ασυλίας του κυρίου Ουσακόφ για να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία για παραβίαση του νόμου διακίνησης στρατηγικών αγαθών. Θα διαβιβαστεί αρμοδίως στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου για τις αποφάσεις ε, των επιτροπών ε, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων δεν έχω κάποιο αίτημα ε, από ομάδες ή βουλευτές ε, το οποίο να ε, επιτυχάνει το κατόφλι. Οπότε μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο πρόεδρος έλαβε από το Συμβούλιο την τοποθέτηση του Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων η προθεσμία των τριών μηνών που έχει το Κοινοβούλιο για να απαντήσει ξεκινάει από αύριο 14 Νοεμβρίου 2020. Πριν ε, ξεκινήσει ο πρώτος γύρος ε, της ε, ψηφοφορίας θα ήθελα να δώσω σύμφωνα με το άρθρο 59 τον λόγο στον κύριο Μπουσόη ο οποίος θα αναφερθεί στο πρόγραμμα EU for Health για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Το έτοιμο αυτό θα τεθεί ε, σε ψηφοφορία. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη χθεσινή ψηφοφορία, για τις τροπολογίες τους και ευχαριστώ όλου του και ηγητές, ε, τον συντονιστή μας ε, Πιτελίζα και όλου του συναδέλφους για την υποστήριξη. Η χθεσινή ε, ψηφοφορία δείξε ότι με 5,1 δισεκατομμύριο το πρόγραμμα όχι θα, δεν θα βοηθήσει μόνο τι μελλοντικέ πανδημίε και τι υγειονομικέ απειλέ, και θα κάνει πιο ανθεκτικό το σύστημα, αλλά θα συμπληρώσει και άλλε πολιτικέ προκειμένου να έχουμε ένα αποθεματικό βασικών φαρμάκων και ε, ιατροτεχνολογικών προϊόντων για καιρού κρίση. Ε, πιστεύω ότι θα, οι διαπραγματεύσει θα είναι επικοδομητικέ και με το Συμβούλιο και θα ολοκληρωθούν πριν τα τέλη του έτου, ώστε το πρόγραμμα να αρχίσει να λειτουργεί ήδη ε, από τον Ιανουάριο του 2021 για να εξυπηρετεί του πολίτε. Οπότε ζητώ παραπομπή στην Επιτροπή για τι διοργανικέ διαπραγματεύσει, άρθρο 59 παράγραφος 4, για το πρόγραμμα EU for Health, Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υγεία. Ευχαριστώ. Περνάμε στην πρώτη σημερινή η ψηφοφορία. Τα θέματα τα οποία ψηφίζουμε αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Η ψηφοφορία είναι από τι 9 μέχρι τι 10 ε, και 4. Θα χρησιμοποιηθεί η ίδια διαδικασία όπω και στου προηγούμενους γύρε. Όλε οι ψηφοφορίε είναι ονομαστικέ. Άρχεται η πρώτη ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι τι 10 και 4. Τα πρώτα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 45. Ευχαριστώ πάρα πολύ.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 Επαναλαμβάνεται η συνειδρίαση και προχωράμε στη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων ε, του πρώτου γύρου ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Ε, μπορείτε να τα διαβάσετε και στην σελίδα. Περνάω στις τελικές ε, ψηφοφορίες. Έκθεση Μπουσόη σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην υγεία εγκρίνεται. Έκθεση Μπουσόη Πρόγραμμα δράσης για την υγεία αναπομπή στην Επιτροπή εγκρίνεται. Έκθεση Μουρεσάν και ΤΑΝΓ Σχέδιο Επενδύσεων ε, για τη Μελλοντική Ευρώπη δεκτό το ψήφισμα στο σύνολό του. Περνάμε στροπολογίες ε, των εκθέσεων Φερνάντες και την Αγγλία... για το πρόγραμμα Invest EU. Διαβάζω τις ε, τροπολογίες. Ένα σημείο β, δεκτή τροπολογία 6, δεκτή αρχικό κείμενο Παράγραφος 1 εδάφιο ε δεκτό. Παράγραφος 7 απορρίπτεται. Τροπολογία 1 CP δεκτή. Τροπολογία 13 καταπίπτει. Η τροπολογία 8 απορρίφθηκε όπως και η 18. Το αρχικό κείμενο άρθρου 5 μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο δεκτά. Τροπολογίες 19 και 20 απερίφθησαν. Αρχικό κείμενο 7 παράγραφος 1 εδάφιο δέλτα μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο δεκτά. Τροπολογία 1 CP μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο επίσης δεκτές. Τροπολογία 1 CP μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο Δεκτές. Τροπολογία 21 απορρίπτεται. Τροπολογία 1 CP. Α, με συγχωρείτε. 21 απορρίπτεται. 1 CP δεκτή. Τροπολογίες 22, 23 και 24 και 25 απερίφθησαν. Τροπολογία 14 απορρίπτεται. Τροπολογία 26 απορρίπτεται. Άρθρο 7, παράγραφος 8, τροπολογία 1 CP δεκτή. Τροπολογία 27 απορρίπτεται. Τροπολογία 4 και 5 απορρίπτονται. Τροπολογία 28, 29 και 30 απερίφθησαν. Αρχικό κείμενο παράρτημο 2 υπαριθμών 13 δεκτό. Τροπολογία 31, 32 δε. 33D, 44D και 35 απερίφθησαν επίσης, όπως και οι 36. Εκτιμώντας 3 οι τροπολογίες 1 CP μέρος πρώτο, 1 CP μέρος δεύτερο και 1 CP τρίτο μέρος έγιναν δεκτές. οι Τροπολογία 15 και 2 επί του εκτιμώντας 10 απερίφθησαν. Η τροπολογία 1 CP για το εκτιμώντας 10 έγινε δεκτή. Για το εκτιμώντας 11. Οι τροπολογίες 9, 3 και 16 απερίφθησαν για το εκτιμώντας 13 οι τροπολογίες 10 και 17 απερίφθησαν για το 24 οι τροπολογίες 1 CP μέρος πρώτο, μέρος δεύτερο, μέρος τρίτο έγιναν δεκτές για το εκτιμώντας 28 οι τροπολογίες 1 CP μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο έγιναν δεκτές για το εκτιμώντας 30. Η τροπολογία 11 απερίφθη. Επίσης, για το εκτιμώντας 30 το 1 CP έγινε δεκτό και η τροπολογία 12 επί το εκτιμώντας 64 απερίφθη. Περνάμε λοιπόν στροπολογίες τροπολογίες για το ψήφισμα επιπτώσεις ε, του COVID-19 στη δημοκρατία, θεμελιώδη δικαιώματα, κράτος δικαίου. Τροπολο... Ε, παράγραφος 3, με συγχωρείτε, τροπολογία 8, απορρίπτεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 2, απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 8, η τροπολογία 18 έγινε δεκτή. Παράγραφος 11, τροπολογία 9, απερίφθη. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 11, μέρος 1 και μέρος 2 έγιναν δεκτά. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 12, έγινε δεκτό. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 14, μέρος 1 και μέρος 2 έγιναν δεκτά. Παράγραφος 15 ή 19 έγινε δεκτή. Αρχικό κείμενο 15 μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο κατέπεσαν. Μετά την 15 ε, απορρίφθηκε η τροπολογία 10 και η 16. Παράγραφος 16 αρχικό κείμενο έγινε δεκτό. Αρχικό κείμενο παραγράφου 17 καταπίπτει άρα. Αρχικό κείμενο στην παράγραφο 19 μέρος πρώτο και δεύτερο έγιναν δεκτά. Αρχικό κείμενο στην παράγραφο 20 μέρος πρώτο μέρος δεύτερο επίσης έγιναν δεκτά. Οι τροπολογίες 11 στην παράγραφο 21 και 12 στην 22 έγιναν, ε, δεν έγιναν δεκτές. Αρχικό κείμενο, αιτιολογική σκέψη 7 έγινε δεκτό. Ε, αιτιολογική παρατήρηση 8, αρχικό κείμενο δεκτό. Αιτιολογική παρατήρηση 9, 12 επίσης δεκτές. Αρχικό κείμενο 13 δεκτό. Αρχικό κείμενο 14 δεκτό. Αρχικό κείμενο 15 δεκτό. Ή θεολογικές παρατηρήσεις 23, 29, 30 και 31 έγιναν επίσης δεκτές. Μετά το εκτιμώντας β απερίφθη η τροπολογία 1 και η τροπολογία 3. Το εκτιμώντας δέλτα 15, 13 ε, με συγχωρείτε απερίφθη. Αρχικό κείμενο εκτιμώντας F μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο έγιναν δεκτά. Τροπολογία 4 έγινε δεκτή. Αρχικό κείμενο τάφ ε, μέρος πρώτο και δεύτερο κατέπεσαν αρχικό κείμενο ΑΑ μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο έγιναν δεκτά. Δεκατέσσερα για τις αιτιολογικές σκέψεις ε, ΑΒ και την τροπολογία 5 επίσης απέριψαν αρχικό κείμενο εκτιμώντας μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο έγιναν επίσης δεκτά. Μετά την αιτιολογική σκέψη ΑΒ απερίφθη η τροπολογία 6, μετά το AC η 15 απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο στο εκτιμώντας AD μέρος πρώτο και δεύτερο έγιναν δεκτά. Αρχικό κείμενο στο εκτιμώντας ΑΕ μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο έγιναν επίσης δεκτά. Τροπολογία 17 έγινε δεκτή και άρα το αρχικό κείμενο AF πρώτος και πρώτο και δεύτερο μέρος καταπίπτουν. Μετά το εκτιμώντας ΑΙ η τροπολογία 7 απορρίπτεται. Άρα μάθατε τώρα όλα τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας και διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 14 Οπότε και θα επανέλθουμε με τον δεύτερο γύρο ψηφοφοριών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας όρεξη. Señor Presidente. Boa tarde. Καλησπέρα σας. λοιπόν τις ε, διαθεσμικές τις διαθεσμικές ε, ε, συμφωνίες όσον αφορά τη δημιουργία του προγράμματος InvestEU και έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Φερνάντες. Θέλω σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου ως εισηγητής αυτού του σημαντικού φακέλου όπου είναι ε, ταυτόχρονα συνεισηγήτρια η κυρία Ιρέν ε, την άλλη. Ήθελα να ζητήσω λοιπόν το InvestEU να παραπεμφθεί στην ε, Επιτροπή Προπολογισμών και Οικονομικών ε, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τις εσωτερικές τις εσωτερικές μας διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να σας συγχαρώ ε, τους συνεισηγητές για την εξαιρετική σας εργασία σε αυτό το θέμα και αυτό το αίτημα θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά από την ψήφιση της πρότασης της Επιτροπής. Και τώρα ξεκινάει η δεύτερη περίοδος ψηφοφοριών για σήμερα. Θα ψηφίσουμε τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια μας διάταξη. Η περίοδος ψηφοφορίας ε, θα ισχύσει ανάμεσα στις 2 και 3 ε, και 4. Η ψηφοφορία γίνεται με την ίδια διαδικασία που έχει ακολουθηθεί στις προηγούμενες περιόδους ψηφοφορίας και όλες οι ψηφοφορίες θα είναι με ονομαστική ψήφο. Αρχίζει λοιπόν η δεύτερη περίοδος ψηφοφορίας για σήμερα. Μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι τις 3 και 4. Τα δε αποτελέσματα αυτής της δεύτερης περίοδου ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν στις 17 ε, και 30, στις 5.30 δηλαδή και για την ώρα διακόπτεται η συνεδρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Επανάληψη τη συνδρίαση και να περάσουμε στα αποτελέσματα της δεύτερης, ε, του δεύτερου γύρου ψηφοφοριών. Τα αποτελέσματα είναι ω εξή. Καταρχά για την έκθεση Φερνάντες και την άλλη για το πρόγραμμα Invest in You. Εγκρίθηκαν την ε, προτάσει το κείμενο δεύτερη έκθεση του κυρίου Φερνάντε και Κινάκη για το πρόγραμμα InvestEU για τις παραπομπέ της Επιτροπές επίση εγκρίθηκε και το ψήφισμα για τι συνέπειε του COVID-19 και σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τα κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Το σύνολο του ψηφίσματος επίση συγκριθήκε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 11ης, 10 και 13ης ε, Νοεμβρίου θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει τα ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν θα χορηγηθούν στα άτομα τα οποία χορηγήθηκαν. Η σύνοδος διακόπτεται. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που συμμετείχαν για την κατανόηση για την συγκεκριμένη κατάσταση η οποία δεν είναι απλή για κανέναν μας. Σας εύχομαι το Σαββατοκύριακο και πέρα στις συνεδρίασεις.